Thank Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Έχουμε πάρα πολλέ ψηφοφορίες, είναι πάρα πολύ μακρύ ο κατάλογο και είναι και πέμπτη και θέλουμε όλοι να γυρίσουμε σπίτι μας. Λοιπόν, όχι πάρα πολλά διαδικαστικά, όσα χρειάζεται και ε, όχι και πολλές συζητήσεις για να τελειώσουμε νωρίτερα.